So, jetzt? Ja. Nochmal alle herzlich willkommen. Ich hoffe... Ελπίζω ότι ξεκουραστήκατε από την πρώτη σειρά των ψυχοφοριών και προχωρούμε τώρα για το 2020. Ο εισηγητής κ. Μπουσόη είναι παρόν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν υποστηρίζει τις συμβαστικές 2 και 3 και η SD 1, 2 και 3. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ή μήπως επιθυμεί ο εισηγητής να λάβει το λόγο. Ναι, σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και ιδιαίτερα την γραμματεία της Επιτροπής ΕΝΒΗ για την ε, σκληρή του δουλειά. Με τις συμβαστικές τροπολογίες ενισχύεται, πιστεύω, η θέση μας στην Ήτρε όσον αφορά τα διάφορα σχέδια της κλιματικές αλλαγές. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε με την ημερήσια διάταξη με το 15 ορίζον 2020. Πρώτη τροπολογία 67 υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, ε, κατά, αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση, 69. Haben Sie alle abgestimmt? Ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 74 υπέρ κάποιος ε, μίλει από κάτω οκ okay, 73 ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει Ψηφίσατε. Πέρασε. 12 υπέρ. 6 κατά. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Καλά, check, οκ. 76 η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Πέρασε. 10 υπέρ, 13 κατά. Απορρίπτεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η ενοποιημένη τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή προχωρούμε στην 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 97 υπέρ θέλετε επαλήθευση επαλήθευση ψηφίσατε όλοι πέρασε 11 υπέρ, 14 κατά απερίφθη. Ε, συγγνώμη, ναι, απερίφθη, καλά το 97 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ψηφίσουμε. 98 λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. 19 υπέρ, 8 κατά και 3 αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 και 103 ταυτόσιμες ψηφίζονται μαζί υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε καλύτερα 100 και 103 ηλεκτρονική επαληθεύση ψηφίσατε Πέρασε. 24 υπέρ 9 κατά εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές αν και νομίζω ότι απορρίπτεται ας κάνουμε την επαλήθευση 105 αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε Τέλος. 20 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. η ψηφοφορία. 22 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά. 116 δεκαέξι, επαναλαμβάνω.

κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117, 119, είναι ίδιες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 115 τώρα. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 125. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στην ενωπημένη της συγκεντρωτική 2. Ο Πίτερ Λίζε. Παρακαλώ. Έχω μία παρατήρηση παρακαλώ να κάνω για την τροπολογία αυτή, την συγκεντρωτική. Ο πρόεδρος και οι συντονιστές πήραν χτες ένα email από τον εισηγητή από την Νομική Επιτροπή. Και το θέμα που τίθεται είναι πολιτικό αλλά και νομικό. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στο mail αυτό. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές απόψεις. Πάντως, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ενέκρινε μία απόφαση που μπορούμε να αγνοήσουμε, αλλά όσοι δεν θέλουν να την αγνοήσουν, πρέπει να πω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταψηφίσουμε τι συγκεντρωτικές τροπολογίες 2 και 3 και να υπερψηφίσουμε την 126. Εννοείται ότι κάνετε ό,τι θέλετε, εγώ απλώς ήθελα να σας το πω να το ξέρετε. Πρόεδρος, ναι, πράγματι πρέπει να αναρωτηθούμε αν ήταν ε, ανάποδα τα πράγματα, αν δίναμε δηλαδή μία ένδειξη εμείς στη νομική επιτροπή, τότε τι feedback, πώς θα έχουμε feedback. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι νιώθω να δεσμεύομαι από αυτά. Ο καθένας μπορεί να υποβάλει τροπολογίες, οπότε ψηφίζουμε τη συγκεντρωτική τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα αλλάξουμε. Συγκεντρωτική τροπολογία 2. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35 υπέρ 20 κατά. Περνάμε τώρα στη συγκεντρωτική 3. Ενωπημένη τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 9. Εδώ δίπλα μου τηλεφωνάνε, εγώ δεν ε, σας ακούω τι λέτε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Α, σας ενοχλώ εσάς που τηλεφωνάτε με ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι της ψηφοφορίας. 56 υπέρ και κανείς κατά. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. 9. Υπέρ. Κατά. Απο... Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158. 139. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 140. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141 υπέρ. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 141. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 37 κατά. Απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Να ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε για την 144 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. πέρα στις ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 49 κατά. Απορρίπτεται βέβαια. 11 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 149, α, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 ε, Ερχόμαστε στα παραρτήματα τώρα. 155 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Α, για την 155 θέλετε να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη 29 29-29 είναι το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. 156 τώρα υπέρ. Κατά. Απο... Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ο, δεν ψηφίζετε όλοι. Οπότε θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 125, 165, συγγνώμη, για την 165 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, πέρα τη ψηφοφορία. 30 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 169 υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 169. Ναι, 168, 168 λέει πρόεδρος. Είμαι σίγουρος ότι έχει περάσει. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Να, το αποτέλεσμα 45 υπέρ, 13 κατά. Σηκώνετε καλά τα χέρια για να σας βλέπω και να μπορώ να μετρήσω τις ψήφους. Αυτό θα μας διευκολύνει όλους. Υπέρ κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 169. Ψηφίσατε όλοι. 31 ψήφοι υπέρ, 28 κατά. Όχι, 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά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 η ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί δεν κατάλαβα το αποτέλεσμα καλά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 50 υπέρ, 9 κατά. Εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. απορρίπτεται, απορρίπτεται, δείχνει ο πρόεδρος. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, εγκρίνεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 221. Υπέρ. Εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φτάσαμε τώρα στη συμβαστική 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στη 228 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 244 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 242 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 238 καταπίπτει. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 241 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 244 ή μάλλον 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 243 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 239 β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 247. Βίλμοτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 254. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 255. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 261 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 262 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 καταπίπτει. 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 έχει αποσυρθεί και φτάνουμε στη 268 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συνεχίζουμε με την 283 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 281 84 και 85 είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 288 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, Θέλετε να επαληθεύσουμε, και εγώ δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για το προηγούμενο 288, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. 39 υπέρ, 21 κατά. Σημαντική διαφορά με αυτά που νομίζαμε. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πηδούμε στην 300 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 301 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 305 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 308 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 310 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 3.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 324 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 325 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 329 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 330 υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 331 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 333 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 334 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.35. Θέλετε 3.34 να επαληθευτεί ηλεκτρονικά. Καλά, αρχίζουμε. Γκέρλινγκ. Εγκρίθηκε λοιπόν 42 υπέρ 19 κατά. υπήρξε σύγχυση γύρω από τα νούμερα και μήπως μπορούμε να ξανακάνουμε την, ε, την ψηφοφορία αυτή, λέει η κυρία Μακάβαν. Πού ακριβώς υπήρξε η σύγχυση. Η μετάφραση του αριθμού στα αγγλικά. Καλά, ψηφίζουμε ξανά ηλεκτρονικά την τροπολογία Julie Gerling με αριθμό 334. Ψηφίσατε. Ψηφίσατε λοιπόν. Ωραία. έληξη η ψηφοφορία. 38 υπέρ, 24 κατά. Παραμένει λοιπόν εγκεκριμένη. 335 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 336 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται αυτή. 3.39 Κοιτάξτε, υπάρχουν και ορισμένοι που διπλοψηφίζουν. Και ναι και όχι. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν την 338, ηλεκτρονικά, 338. 338 ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. 25 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. 339 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 347 όχι ακούγονται φωνές επανάληψη Καλά λοιπόν, 346 ηλεκτρονική υπολήθευση. Ψηφίσατε. Τέλος. 45 υπέρ, 15 κατά. Κανένα, καμία δυνατότητα να το δω από εδώ ψηλά. 347 υπέρ. Α, ναι, εκπίπτει, εκπίπτει, σωστά. 348 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβατική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και στην, πηγαίνουμε 353, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 355, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 356, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 350, όχι, 8, 358 ναι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 359 υπέρ. Ε, κατά αποχές απορρίπτεται. 360 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 361 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 367 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 368 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 381 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 382 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 383 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 384 υπέρ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 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές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 μία ψήφος κατά και δέκα αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Παραμένουμε στον ίδιο εισηγητή και προχωρούμε στο πρόγραμμά μας με το 17, δηλαδή την εφαρμογή του Horizon 2020 και με πρώτη τροπολογία που τίθεται σε ψηφοφορία την 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ. Α, καλά, θα επαληθεύσουμε την 58. Ναι, ναι, οκ. Okay. Έλεγχος. Ψηφίσατε και βλέπω ότι ήταν μεγάλη πλειοψηφία, 45 υπέρ 13 κατά και καμία αποχή.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 αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. <coughs> Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ.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 κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Επαλήθευση της 85 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 17 υπέρ και 44 κατά. Καθαρή απόρριψη.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 κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλύτερα να επαληθεύσουμε όμως. Την 104. Ψηφίσατε. Τέλος. Βεβαίως. 54 υπέρ, 7 κατά. 102 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120 υπέρ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 εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 121 λέει ο πρόεδρο, αλλά νομίζουμε ότι εννοεί 21. 21 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται και αυτή. Πηγαίνουμε τώρα στην Consolidated 5, ενωπημένη 5, υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά θα προβούμε σε επαλήθευση 144 ηλεκτρονικά ψηφίσατε πέρασε 31 ψήφι υπέρ 30 κατά είναι λοιπόν θετική η ψήφος 146 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 146 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Τέλος. 32 υπέρ, 28 κατά και μια αποχή. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 148 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 <coughs> συγγνώμη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επαληθεύουμε όμως την 169 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Τέλος ψηφοφορίας. 29 ψήφι υπέρ, 31 ψήφι κατά. Απορρίφθηκε. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά ψηφίσατε παρακαλώ όλες και όλοι τέλος της ψηφοφορίας ψήφι 36 υπέρ 26 κατά 177 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται και αυτό. 181 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 3... 132 λέει ο πρόεδρος, 32 ίσως εννοεί. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά.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 Λοιπόν, να το ελέγξουμε. Δεν είναι προφανές. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 59 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί του συνόλου. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 62 υπέρ. Κανείς κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Για την ε, σκληρή δουλειά. Τώρα στο αγαπημένο μας πρόγραμμα. Life. Ε, λοιπόν, πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία, να έχετε υπόψη σας ότι τροπολογίες 36 ε, ορισμένες τροπολογίες δεν είναι αποδεκτές διότι έτσι αποφάσισε το Προεδρείο. Και οι 89 και 90 αποσύρθηκαν. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Ρεγγί 12 υπέρ. κατά αποχές ωραία θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο όχι έχει αρχίσει η ψηφοφορία δεν ζητήσατε την αρχή ψηφοφορία ζητήσατε κατά τη διάρκεια αγαπητέ συνάδελφοι έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Όσο και να φωνάζετε δεν αλλάζει τίποτα. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Μετά θα πάρετε το λόγο για το διαδικαστικό. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 υπέρ, 20 κατά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. είχα την ευκαιρία να στείλω ένα μήνυμα σε σχέση με την ε, απόφαση να μην γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες 63, 64 και 65. Κατά τη γνώμη μου, όπως θα είδατε και σε αυτό το μήνυμα, η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη και δεν έχει καμία βάση, ακόμα και υπό το φως ε, της απόφασης ε, του Προεδρία. Η τροπολογία 65, της οποίας είμαι εγώ συντάκτης και που έχει το ίδιο νόημα με τις 63 και 64, δεν προτείνει συγκεκριμένα ποσά όσον αφορά τον προπολογισμό. Αυτό είναι το αμφισβητήσιμο και αυτό είναι που η απόφαση αφορά. Ότι δηλαδή να μην κάνουμε προτάσεις με, καμία συγκεκριμένο, με κανένα συγκεκριμένο νούμερο. Απλώς πρόκειται για επιβεβαίωση μιας πολιτικής αρχής όπου με βάση την οποία θεωρούμε ότι ανεξάρτητα με το ποιοι θα είναι οι πόροι που θα δοθούν ε, μέσα στο πλαίσιο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να πάρει το 1% του προπολογισμού. Δεν μιλάμε δηλαδή για νούμερα εδώ, δεν μιλάμε για, μιλάμε για μια αρχή πολιτική. Δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να ψηφίσουμε ε, σε αυτή την Επιτροπή, η οποία είναι κυρίαρχη. Μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να ψηφίσει υπέρ ή κατά. Τώρα να μην δεχτείτε καν τις τροπολογίες αυτές ε, είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μας. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Η διάσκεψη των Προέδρων και η διαπραγματευτική ομάδα και στην Επιτροπή Προπολογισμών. Όλοι αυτοί αποφάσισαν και με μεγάλη πλειοψηφία ότι δεν θα αναφέρουμε συγκεκριμένα ποσά και ούτε ποσοστά. Διότι είμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Να το σεβαστούμε. Ε, Αλλιώ απευθυνθείτε σε αυτά τα όργανα που πήραν αυτέ τι αποφάσει. Εγώ ακολουθώ αυτή τη γραμμή που συμφωνήθηκε μεταξύ των διαφόρων οργάνων του σώματος. Και περνάμε λοιπόν στο τροπολογία 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 συνολική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, να το ελέγξουμε. 89, ηλεκτρονικός. Άρχεται. Πέρασε. 34 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 με μια προφορική προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ όχι καλά να ελέγξουμε την 90 Κανένα πρόβλημα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 36 υπέρ. 24 κατά. Εγκρίνεται. Παρακαλώ ε, ε, να σηκώνετε τα χέρια σας. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μετρήσω αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας και μόνο με το κεφάλι άμα κάνετε. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε μπορούμε να πάμε αρκετά παρακάτω. Ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε, τροπολογία 106 και 107. Α, καταπίπτουν, καταπίπτουν. Α. Εκατόν εξήντα υπέρ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 167 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 167 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 19 υπέρ, 38 κατά. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπουτζ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 34 και ίτρε 10 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 123 124 και Ρέγγι 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Οκ, okay, να ελέγξουμε. Τις τρεις τροπολογίες 123, 124 και 17 ηλεκτρονικός. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 37 υπέρ 24 ε, κατά εγκρίνονται. 125 και 126. Δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε. Οπότε περνάμε στην 35 και ρέγγι 16. Λέει ο πρόεδρος. 19. Ρέγγι 19 Διόρθωνα ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 36 και ήτρε 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ήτρε 14 υπέρ. Ήτρε 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 14 υπέρ. Κατά αποχές ασαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. Ήτρε 15 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 και ρέγγι 20 ταυτόσιμες. Από κοινού υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ρέγγι 21 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 129 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε 133 ψηφίσατε όλοι πέρασε 31-30. Εγκρίνεται. Ενωπημένη 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 27. Υπέρ κατά αποχές κρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέγγι 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 141 ψηφίσατε όλοι πέρασε 30 προς 31 απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 144 και ρέγγι 31 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 44 και 145 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ενοποιημένη 4β υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκριν... Απορρίπτεται η 4β, λοιπόν, ενοποιημένη. Ενοποιημένη 4α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλά, ελέγχουμε. 4α. Σιγουριά καλύτερη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 33 με 28 εγκρίνεται. Ενοποιημένη 4 σε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Wir kommen jetzt zum Abänderungsantrag 165 τώρα παρακαλώ. Περνάμε στην 165. Ποιοι είναι υπέρ. Ε, εγώ έχω στη σελίδα 14 165, αλλά δεν ξέρω αν ο, ο κατάλογος του Έλκη είναι ο ίδιος. Λοιπόν, 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 170 με μία προφορική προσθήκη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε την αρχική 170 χωρίς προφορική προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ της ε, αρχικής 170. Επαναλαμβάνω ποιοι είναι υπέρ της 170 στην αρχική της μορφή, χωρίς την προφορική προσθήκη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενοποιημένοι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλά, καλά να ελέγξουμε. Ευχαρίστως. ηλεκτρονικά την ενοποιημένη 5. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 39 υπέρ, 21 κατά. Και μία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Κατά αποχές εγκρίνεται. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Η τροπολογία 165 κατά τη γνώμη μου δεν είναι σύμβατη με τη συμβαστική 5 που μόλις εγκρίθηκε. Κρίνω πως αυτή η τροπολογία μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη στην συμβαστική 5. Η 100 75, με συγχωρείτε, ε, αφορά το, τα ποσοστά ε, και των μέτρων που όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί. Η 5 δε αναφέρεται στις ε, περιφέρειες με συγκεκριμένες προτεραιότητες. Δεν είναι ασύμβατη λοιπόν αυτή η τροπολογία με τη συμβιβαστική και γι' αυτό πρέπει να την ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε όπως συμφωνήθηκε με τις ομάδες. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τον κατάλογο ψηφοφοριών. Συμβαστική 7. Υπέρ. Α, είχαμε ψηφίσει, είχαμε ψηφίσει. Δεν είχαμε ψηφίσει. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189-90 έχουν αποσυρθεί. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 192 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 προς 36 απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 με προφορική προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 36 και 196 ταυτόσημες κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 με μια προφορική προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 και 21 ήτρα ίδιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρα 22 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Ωραία. Έλεγχος 200, 22 ε, Ήτρε. Ήτρε 22. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22-35. Απορρίπτεται. Ήτρε 22. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενωπημένη είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε, τροπολογία, badge 5, στη σελίδα 24, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Budget 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 και Ρέγγι 2 ταυτόσιμες από κοινού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ήτρε 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 3 υπέρ. Κατά αποχές Να το ελέγξουμε, να το ελέγξουμε. Ρέγγι 3. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Μάλιστα. Σαφές. Σαφής απόρριψη. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέγγι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπάτζο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 και ρέγγι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 με μια προφορική προσφυγική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 79 έχει ήδη εγκριθεί, οπότε πάμε 14, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ή 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενωπημένη 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε. Τελική ψηφοφορία όπως πάντα, ηλεκτρονικός για το σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 56-2-2. Οπότε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 56, 3, 1. Μία. Συγχαρητήρια στη Utah Hawk. Νομίζω ότι είναι ορόσημο αυτό για το πρόγραμμα Live, για το περιβάλλον στην Ευρώπη. Συγχαίρω ιδιαίτερος και ευχαριστώ πολύ για την πειθαρχία που επιδείξατε κατά την ψηφοφορία. Ξέρω ότι σήμερα ε, χρειάστηκε να εργαστούμε πολύ. Όσοι θέλουν να μείνουν, χαίρομαι που θα μείνουν. Όσοι θέλουν να φύγουν, θα τους παρακαλούσα να φύγουν τώρα. Σας παρακαλώ, όσοι επιθυμούν να παραμείνουν, να καθίσουν πάλι στις θέσεις τους και όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα μπορούν βεβαίω να το κάνουν για να συνεχίσουμε. Κάπως μας πιέζει ο χρόνος και εγώ θέλω να δώσω τον λόγο στον εισηγητή κύριο Σνέλχαρτ. Gut, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Πολλοί φεύγουν και φαίνεται πως δεν έχουν κατοικίδια και δεν ενδιαφέρονται να τα πάρουν μαζί τους σε ταξίδια. Βέβαια εγώ ούτε έναν βουλευτή δεν έχω δει σε όλη τη διάρκεια που επεξεργάζομαι την έκθεση να έρχεται εδώ με συνοδεία κάποιου κατοικίδιου, ίσως και να μην επιτρέπεται. Πάντως τώρα για την έκθεση που έχουμε μπροστά μας, πρόκειται για τα καταλήματα, κατοικιδίων, βεβαίως και για εμπορικούς ε, λόγους, εφόσον δηλαδή η οικογένεια Σμιτ παίρνει το σκυλάκι της και πηγαίνει σε άλλη χώρα, πώς αυτό θα γίνει. Αυτό συζητείται και ε, σχολιάζεται στην έκθεση. Μπορείτε να τα διαβάσετε βεβαίω αυτά. Θα θυμάστε ότι προδιετίας νομίζω είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ιδιαίτερε ρυθμίσει για τη Μεγάλη Βρετανία και τις σκανδιναβικέ χώρες να σταματήσουν να ισχύουν, διότι δεν υπήρχε πλέον βάση για αυτές. Αυτό ζητείται λοιπόν τώρα και ρυθμίζεται μάλλον στην πρόταση της Κομισιόν. Εξού και η νέα αλλαγή και η τροποποίηση της εκθέσεως που καθίσταται απαραίτητη για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις στη συνθήκη της Λισαβόνας. Με μεταβατική περίοδο ο χαρακτηρισμός των ζώων και άλλες σχετικές διατάξεις. Αυτές είναι οι βάσεις για τις τροποποιήσεις αυτές του κανονισμού που αποτελείται από δύο βασικά κεφάλαια αφενός τους όρους για την εισαγωγή κατοικιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για την διακίνηση κατοικιδίων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης χώρας. Και μιλεί εδώ για γάτους, σκύλους και νηφίτσες. Καθώς επίσης με ειδικέ ρυθμίσεις για πολύ νεαρά ζώα και ορισμένες εξαιρέσεις. Πρόκειται και για μέτρα προληπτικά εξασφάλιση της υγείας των ζώων, για ταυτότητες των κατοικιδίων, που ε, είναι έγγραφα τα οποία οφείλουν να συνοδεύουν το ζώο. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν. στόχος είναι και για μένα και για την Κομισιόν να διευκολυνθεί η μετακίνηση με συνοδεία κατοικιδίων χωρίς να υπάρξουν προβλήματα ή κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Εγώ προσπάθησα να κάνω την έκθεση πιο ευνόητη, πιο ευανάγνωστη. Αυτό οδήγησε βέβαια σε ένα αριθμό τροπολογιών που δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε σύγχυση, διότι πάμε να άρουμε μία ρύθμιση της Κομισιόν και να την καταστήσουμε με άλλη. Γίνεται λοιπόν αρκετά εκτεταμένη έκθεση, αλλά θεώρησα ότι αυτό είναι απαραίτητο, διότι ιδίω για θέματα ταυτότητων ε, των ε, ε, ζώων πρέπει να περιέχονται ορισμένα στοιχεία και αυτά είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν. Ζητούμε εμείς λοιπόν πολύ συγκεκριμένες και λεπτομερείς ρυθμίσεις, να υπογράψει δηλαδή και ο ιδιοκτήτης και ο κτηνίατρος και οι δημόσιες αρχές θα ορίσουν ποιος κτηνίατρος επιτρέπεται να το κάνει και όχι. Έχουν υπάρξει πολλές ανομαλίε τον ε, τελευταίο καιρό όπου πολλοί προσπάθησαν να πλαστογραφήσουν τις ε, ε, άδειε αυτές, τι ταυτότητε αυτές. Οι βασικές προϋποθέσεις για το τι θα διαλαμβάνουν αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονται στον κανονισμό πλέον. Σε ένα θέμα ξεφεύγω λίγο από την πρόταση της Κομισιόν. Έχω λάβει πολλές επιστολές από διαφόρους οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινήσουν σκυλιά τα οποία τραβούν έλκυθρα. Και εκεί αντιμετωπίζουν τον περιορισμό των πέντε κατοικιδίων, οι πέντε ζώων που έχει προτείνει ανά πρόσωπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έχουν τότε προβλήματα για να διαβούν τα σύνορα και δεν μπορούν να συμμετάσχουν τότε στους σχετικούς αγώνες. Προτείνω στην έκθεση αυτή να καταστεί δυνατή αύξηση του αριθμού αυτού υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι προποθέσει θα πρέπει να είναι ότι κανείς οφείλει να αποδείξει ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε αθλητική ή άλλη σχετική εκδήλωση. Ότι συμμετέχει σε κάποιον όμιλο ή ε, σύνδεσμο. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε ένα κενό της οδηγίας που είχε μέχρι τώρα που προκαλούσε προβλήματα που χρειάζονταν ειδικέ άδειε και ούτω καθεξής από τις ε, ε, αρμόδιες αρχές. Αυτό λοιπόν εδώ τώρα έχει εξαλειφθεί. Υπήρχε και μια θεά ζώνη για τους μη, για τους μη ειδικούς. Υπάρχει το θέμα των εμβολιασμών. Κάθε ζώο το οποίο μετακινείται στο εξωτερικό πρέπει να είναι εμβολιασμένο, ίσχυε μέχρι τώρα και ισχύει ακόμη, αλλά για ζώα ηλικίας από 0 έως 12 μηνών έχουν και κάποια προστασία από την ε, μητέρα, αλλά μετά τους 12 μήνες πρέπει να εμβολιάζονται. Δεν θα πρέπει να μετακινούνται τότε στο εξωτερικό, στην Αλοδαπή. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να μπορούν να συνοδεύουν τα φοιτικά τους στο εξωτερικό. Τώρα, νομίζω ότι έχει ρυθμιστεί αυτό, διότι περιλάβαμε το θέμα αυτό και είπαμε ακριβώς αυτά τα ζώα μπορούν και αυτά να πηγαίνουν με την πλήρωση ορισμένων όρων, δηλαδή να μην έχουν έλθει σε επαφή με ζώα τα οποία ίσως αποτελούν κίνδυνο μόλυνσης. Νομίζω ότι γενικά έχουμε επιτύχει διευκόλυνση υπέρ των πολιτών μας και ταυτόχρονα πλέον συγκεκριμένη, πλέον ακριβή διατύπωση για το περιεχόμενο των ταυτοτήτων που συνοδεύουν τα κατοικίδια. Και νομίζω ότι έτσι κάναμε μια σημαντική πρόοδο και εξασφαλίζουμε καλύτερη ρύθμιση. Η δεύτερη έκθεση αναφέρεται σε εμπόριο ζώο, ζώων, σε ζώα που είναι αντικείμενο εμπορίου, είτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τρίτε χώρε. Εδώ δεν έχω αλλάξει τίποτα στην πρόταση τη Κομισιόν, διότι η πρόταση τη Κομισιόν προβλέπει πολύ περιορισμένε αλλαγέ. Μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε ήταν ότι η απόδειξη της, της υγειονομικής εξέτασης του ζώου έπρεπε να είναι πρόσφατη, μέχρι σε 24 ώρες πριν από την διάθεση του εμπόριου. Φάνηκε όμως στην πράξη ότι ήταν υπερβολικά βραχυπρόθεσμο αυτό. Και υπάρχουν και άλλες διεθνείς διατάξεις που λένε 48 ώρες. Δεν έχω κάποια αντίθεση λοιπόν, το βρίσκω ε, σωστό γιατί επιφέρει και μια διευκόλυνση χωρίς ε, στην πραγματικότητα να χαλαρώνει τις ε, προβλέψεις για την προστασία της υγείας. Και μπορεί να μπει και στον κανονισμό για τις μεταφορές που έχει ψηφιστεί και στο Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι μπορούμε να δηλώσουμε ικανοποιημένοι. Δεν έχω λοιπόν προβλέψει άλλες τροποποίησεις για την, στην έκθεση αυτή μάλλον και αναμένω βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Σνέρχαρτ. Πρόκειται για τα θέματα 21 και 22, 22 της ημερησίας τα οποία συζητούνται μαζί. Θα ακολουθήσουν οι σκιώδεις συζητητές. Πρώτος ο κύριος Γιούστας Παλέτσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι, πιστεύω, να είναι εύκολα κατανοητός ο κανονισμός όχι μόνο για τους επαγγελματίες, τους κτηνίατρους δηλαδή, αλλά και για τους απλούς ιδιοκτήτες κατοικιδίων. Ε, πιστεύω πως οι προτάσεις του εισηγητή είναι σωστές. Μόνο και μόνο ο όγκος των τροπολογιών, κύριε Σνέλχαρτ, που κάνατε, 160 τον αριθμό, δείχνουν ότι αφιερώσατε πολύ χρόνο στην υπόθεση αυτή και καταφέρατε να φτιάξετε ένα έγγραφο που είναι που να μιλά στους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες. Σύμφωνο με το ότι το μοντέλο ενός ε, είδους ταυτότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό και θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η προστασία αυτών των εγγράφων από πλαστογράφηση. Η προτινόμενη εξαίρεση ότι πάνω από πέντε ε, ζώα μπορούν να συνοδεύουν ε, τον ιδιοκτήτη, αν ο ιδιοκτήτης ε, μεταβαίνει σε κάποια έκθεση, σε κάποια αθλητικό, αθλητική εκδήλωση, είναι αποδεκτή. Όμως θα πρέπει να υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες για να μην γίνεται κατάχρηση αυτής της εξαίρεσης. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι να ζητήσουμε ηλεκτρονική ε, γραφή ε, online για τα συγκεκριμένα, ζώα. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων ε, πανευρωπαϊκή. Θα είναι έτσι δυνατόν να πάρουμε πληροφορίες για τα κατοικίδια ενός κράτους μέλους, να επαληθεύουμε τον ιδιοκτήτη του και άλλες σχετικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σνέλχαρτ. Δεν έχω ακούσει καμιά επίκριση για την έκθεσή σας. Η κατεύθυνση την οποία ακολουθείτε είναι ρεαλιστική και λογική. Μόνο επένους ακούω όσον αφορά τις προσπάθειές σας για απλοποίηση της διατύπωσης. Ένα-δύο ερωτήματα εγώ έχω στο μυαλό μου. Το ένα είναι κατά πόσο η απόδειξη που θα χρειαστεί, για παράδειγμα όταν κανείς μπαίνει σε ένα κατάστημα κατοικιδίων, αν ε, αυτό θα ε, αρκούσε για να αιτιολογηθούν οι εξαιρέσεις που προτείνονται. Μήπως δηλαδή πρόκειται για κάποιο εμπόριο που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη εξαίρεση και να δώσει ψευδείς ε, ταυτότητες. Ένα ερωτηματικό έχω εκεί και θα προσπαθήσω να βρω κάποιες απαντήσεις για αυτές τις ε, ανησυχίες. Και έπειτα έχω κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσο σε ε, ορισμένα σημεία οι προτάσεις για κεντρικά Μητρώα, μήπως είναι κάπως υπερβολική, πολύ ρύθμιση και νομοθεσία. Όμως τα κράτη-μέλη είπαν ότι θα ήταν λογική βελτίωση. Θα ήθελα ωστόσο να το σκεφτώ τις επόμενες εβδομάδες και να το διερευνήσω να δω αν υπάρχουν σχόλια σχετικά με αυτό. Αλλά με πολύ ενδιαφέρον περιμένω τα όσα έχει να μας πει η Κομισιόν σε σχέση με αυτήν την έκθεση και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε, Κρίς Davis. Η είναι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί κόσμος ε, και όπως και εγώ ταξιδεύουμε με κατοικίδια ζώα και ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει κανείς να έχει μαζί του, ποια είναι τα εμβόλια που πρέπει να έχει κάνει για να μπορέσει να πάρει μαζί του το τετράποδο φίλο του. Είναι αλήθεια ωστόσο ότι τα περισσότερα τετράποδα ή κατοικίδια δεν περνούν τα σύνορα τόσο συχνά, πολλές φορές ποτέ στη ζωή τους και δεν θα ήθελα αυτός ο κανονισμός να επιβαρύνει ένα σωρό κόσμο που δεν ενδιαφέρεται. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου ήδη ισχύουν ένα σωρό μέτρα μικροτσίπ, συγκεκριμένα ε, σημάδια στα αυτιά των ζώων κτλ. κτλ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. που βελτιώνει μάλιστα την πρόταση της Κομισιόν. Η ομάδα μας θεωρεί πως είναι σημαντικό να γίνουν αλλαγές που θα περιορίζουν τις υπερβολικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Ε, να δοθεί δηλαδή για παράδειγμα μεγαλύτερη ευελιξία στα κρατημέλη ώστε να μπορούν να καθορίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται. Και θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε από τον εισηγητή Ποιε είναι οι πιο συγκεκριμένε του προθέσει όσον αφορά κάποιε πτυχέ. Οι προτάσει τροπολογιών όσον αφορά τη διαδικασία microchip θα θέλαμε να μας εξηγηθούν κάπως καλύτερα με περισσότερες λεπτομέρειες από τον εισηγητή. Και υπάρχει και ένα θέμα αρμοδιότητας όσον αφορά την ρύθμιση για τα μικροτσίπ που καθορίζει, που σημαίνει μάλλον εμπλοκή και των τοπικών αρχών. Και το συγκεκριμένο θέμα θα αποτελέσει επιπλέον φόρτο για τις τοπικές αρχές. Το σημείο κίνησης είναι σωστό όμως και γι' αυτό ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κοιτάξτε, είναι πολύ καλό να μπορεί κανείς να μεταφέρει τα κατοικίδια ζώα του διασυνοριακά έχει ιδιαίτερα δοθεί έμφαση στην λύσα, στην ασθένεια αυτή και υπάρχουν και κάποιο είδους ε, ασθένειες που προκαλούνται από σκουλίκια, τα οποία είναι παράσιτα και ζουν στα έντερα των ζώων. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, ε, υπάρχει μεγάλη κουβέντα όσον αφορά ε, τη, τα, τα, τα κατοικίδια ζώα και το κατά πόσο αυτά μπορεί να μολύνουν το μέρος όπου κατοικούν και τους ανθρώπους. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις Πράγμα το οποίο νομίζω μπορεί να, να, να δημιουργήσει πρόβλημα. Ας πούμε και εμείς όταν πάμε να μαζέψουμε ε, καρπούς στο δάσος μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για προσβρώση Πολύ καλό λοιπόν να δημιουργηθούν κανόνες για το πέρασμα των συνόρων για τα ζώα, αλλά και οι χώρες οι οποίες ακόμα δεν έχουν αυτά τα παράσιτα να μένουν ανέπαφες, γιατί διαφορετικά ε, πρόκειται για πολλά δισεκατομμύρια όσον αφορά τις ζημιές που θα πάθουν οι χώρες αυτές αν περάσουν τα παράσιτα. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν κάποιες απαιτήσει όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σλίτερ, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, που είναι ο τμήματάρχη της Γενικής Διεύθυνσης ε, Υγείας και, κατανο... και Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδεξη με την έννοια ότι στόχο έχει να αποσαφηνίσει έναν τομέα και έναν κανονισμό που δεν είναι πολύ σαφής σε ορισμένες του και μάλιστα θεωρείται πια ξεπερασμένος υπό το φως της ηθίκης της Λισαβόνας. Γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει στόχο να εισάγει ριζικές αλλαγές για έναν κανονισμό που θεωρούμε ότι έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής αρκετά καλά. Αν σκεφτούμε ότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια που υιοθετήθηκε, υπήρξε αντικείμενο μακρών συζητήσεων και δύσκολη συμβιβαστική λύση, μπορούμε ωστόσο να πούμε πω τα πράγματα δέκα χρόνια μετά λειτουργούν σίγουρα καλύτερα και η προσυκανοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών που μπορούν να έχουν τη χαρά να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδια του ζώα με ασφαλή τρόπο αλλά και χωρί μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο. Γι' αυτό και η πρόταση τη Κομισιόν Φυσικά προσπαθεί να ξεκαθαρίσει όσο γίνεται και να απλοποιήσει τους ισχύοντες κανόνες, να τους προσαρμόσει και μάλλον να τους προσαρμόσει στη συνθήκη της Λισαβόνας. Φυσικά μας χαροποιεί όλη η δουλειά που έκανε ο εισηγητής κ. Σνέλχαρτ που ακριβώς αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί, δηλαδή να συμβάλλει εν τέλει σε μια βελτίωση και όσο γίνεται και σε μια απλοποίηση των κανόνων. Είναι κανόνες που είναι άμεσα εφαρμοστέοι για εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που ταξιδεύουν με τα κατοικίδια τους ζώα. Γι' αυτό και λάβαμε με χαρά το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Σνέλχαρτ που περιλαμβάνει ένα σωρό ε, ε, παρατηρήσεις πολύ κέρυες με χαρά επίση θα συνεργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες με το Κοινοβούλιο ώστε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την πρόταση της Κομισιόν. σα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Να ξαναδώ το λόγο στον εισηγητή, κύριε Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις ε, προτάσεις, τη συζήτηση. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την ε, θέση της. Συνάδελφοι, για τα πλαστά έγγραφα, κύριε Ντέβις. Η πρότασή μα ε, θα καθιστά σχεδόν αδύνατο να υπάρχουν τέτοια παραχαραγμένα έγγραφα, διότι θα υπάρχει σύγκριση των εγγράφων τους ώστε να είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει ε, παραχάραξη προς την κυρία Ρόσμπαχ. Νομίζω ότι χρειάζονται αυτές οι διατάξει. Ο κύριο Λίτερ είπε ότι η κατάσταση σε ορισμένε χώρες είναι διαφορετική. Πρέπει να έχουμε μια συνολική εποπτεία και έλεγχο, ούτω ώστε να μην αλλάξει κατάσταση σε κάποια περιοχή και αυτό να οδηγήσει σε νέες καταστάσεις δυσάρεστες. Είναι σημαντικό αυτό. Ήδη στον κανονισμό έχουμε ότι η σήμανση θα γίνεται με ένα μικρό τσίπ. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες μήπως κάποιοι δεν μπορούν να το διαβάσουν σε άλλες χώρες. Μπορούν να συνεχίσουν και τα άλλα σημάδια σήμανσης. όσες έχουν υπάρξει πριν την 3η Ιουλίου 2011 και βεβαίως θα πρέπει να μπορεί αυτό το microchip, microchip να αναγνωρίζεται για να υπάρχει ταυτοποίηση του ζώου. Τέθηκε το θέμα της τράπεζας δεδομένων, του Μητρώου. Ξέρω ότι πολλοί στο Κοινοβούλιο που ασχολούνται με το θέμα αυτό μου έθεσαν το θέμα εάν πρέπει να υπάρξει μία τράπεζα σε πανευρωπαϊκό δεδομένο. Αν ε, ο στόχος μας είναι να εμποδίσουμε να υπάρχουν αδέσποτα ζώα. Κάτι που δεν θα το εμποδίσουμε νομίζω. Ή αν χαθεί κάποιο ζώο να μπορούμε να το ξαναβρούμε. Δεν είναι ρεαλιστικές αυτές οι φιλοδοξίες. Αυτό θα σήμαινε ότι οποιοδήποτε έχει μια γάτα να βάλει ένα τσίπ στη γάτα του και να το δηλώσει στην τράπεζα δεδομένων. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό. Δεν είναι αναγκαίο δεν μας φέρνει καμία ασφάλεια. Βεβαίως θα κερδίσουν πολλοί όσοι θα διαχειρίζονται αυτές τις τράπεζες δεδομένων. Δεν θα είναι ούτε θελοντικό αυτό, ούτε χωρίς κόστος. Είναι υπερβολικά όλα αυτά. Πριν από δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο μιλήσαμε για τη σήμανση των βοηδών πρέπει να υπάρχει ε, σαφής σήμανση του ζώου και εγγραφή για να έχουμε μια συνολική εποπτεία ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ζώου. Αλλά τώρα να υποχρεώσουμε τους πάντες να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Όποιος θέλει να εγγράψει το ζώο του μπορεί να το κάνει ιδιωτικός και αυτό μετά θα μεταφερθεί και θα είναι παντού ανακοινώσιμο. Νομίζω θα ήταν υπερβολικό αν θέλαμε αυτό να το βάλουμε στο νομοθέτημα. Παρακαλώ τους συναδέλφους να το ξανασκεφτούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Σνέρχαρτ. Chris Davis, πολύ σύντομη παρέμβαση. Ερώτηση προς εισηγητή ή κομισιόν. Δέκα χρόνια είπατε έχουν περάσει από την πρώτη εισαγωγή αυτή της ρύθμισης για την διακίνηση γάτων, σκύλων και νηφιτσών. Έχουμε καθόλου νούμερα για το πόσες τέτοιες διακινήσεις έχει, ε, έχουν υπάρξει. Ο εγώ προτιμώ να διαβιβάζω την ερώτησή σας κατευθείαν στην Κομισιόν, διότι δεν μπορώ να γνωρίζω το εμπόριο βέβαια σίγουρα είναι σημαντικά τα νούμερα. Αλλά γνωρίζω ότι ορισμένοι πολίτε παίρνουν μαζί τα ζώα συντροφιά και αυτού καλύπτει αυτή η ρύθμιση που συζητούμε τώρα. Όμω, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μεταφέρετε την ερώτηση περαιτέρω προ την Κομισιόν, ίσω γνωρίζει περισσότερα. Βέβαια, εάν ούτε η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει, τότε εγώ θα ψάξω να βρω τα νούμερα αυτά. Φαίνεται πως ο Chris Davis πέτυχε τον στόχο, τον στόχο του ακριβώς, διότι βλέπω ότι άλλα χέρια κατέβηκαν. Η κυρία Ρόσπαχ. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ έχω δύο θέματα. Άκουσα πρόσφατα από τον κύριο Σνερχάρτ ότι δεν θα μπορούν όλοι οι κτηνίατροι να εκδίδουν τις ταυτότητες αυτές. Αυτό είναι μόνο γερμανική ρύθμιση. Και η δεύτερη ερώτηση. Ακούω από την δανική αστυνομία ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτά τα τατουάζ. Διότι κάθε φορά που βρίσκουν μια σκοτωμένη γάτα στο δρόμο δεν έχουν ε, το ειδικό νηστέρι που επιτρέπει την αφαίρεση του τσίπ για να μπορέσουν μετά να το διαβάσουν κτλ. Καλά, εδώ θα κλείσω όμω τον κατάλογο των αγορητών. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο ε, Σνέλχαρτ και μετά θα απαντήσει η Κομισιόν. Ναι, κοιτάξτε, Πώς ήταν η πρώτη ερώτηση. Καλά, μου την ξαναλέτε. Για τη δεύτερη, για αυτό το τσίπ Πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια ενιαία ρύθμιση. Η γάτα, η οποία, κοίτα, ή μάλλον ανεβρίσκεται στο δρόμο, τη βρίσκει κάποιο δρόμο, μάλλον συνήθω δεν έχει chip. Το chip αυτό δεν είναι υποχρεωτικό γενικά για όλα τα ζώα στην Ευρώπη. Μόνο εφόσον κάποιο θέλει να μεταφέρει το, το ζώο συντροφιά εκτό χώρα. Υπάρχει ρύθμιση σε ορισμένε ε, χώρε μέλη, βέβαια δεν είναι μόνο η γερμανική ρύθμιση αυτή. Α, ναι, η πρώτη ερώτησή σα ήταν σχετικά με τον κτηνίατρο. Είναι μια νεοϊσαχτής αρρύθμιση αυτή, όπου βέβαια η αρμόδια αρχή καθορίζει ποιοι κτηνίατροι επιτρέπεται να εκδίδουν τι αδείε αυτέ. Εγώ υποθέτω ότι θα είναι αρκετά ευρύ ο κύκλο των προσώπων αυτών που θα λάβουν τη σχετική άδεια αλλά κάποια εποπτεία πρέπει να έχουμε, διότι ακριβώς τον τελευταίο καιρό σημειώθηκαν πολλές νοθεύσεις. Κάπως πρέπει να μπει κάποια τάξη και να μπει μια ιεραρχία έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι απόπειρες πλαστογράφησης ή νόθευσης και τα ζώα αυτά τελικά να περνούν έτσι καταχρηστικά στο εμπόριο. Να μπορούμε λοιπόν να υπάρχει μια ιχνηλασιμότητα, να μπορούμε να βρούμε ποιο εξέδωσε το σχετικό έγγραφο και το καθεξής. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, σύντομα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Όσον αφορά τις στατιστικές, δεν έχουμε αυτή είναι αλήθεια. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η Κομισιόν δεν μπορεί να, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ένα αυτοκίνητο ε, που πάει από, τακτικά από το Βέλγιο στο Λουξεμβούργο έχει και ένα σκύλο μέσα και αν σε μισή ώρα θα πάει και στη Γαλλία. Τέτοιου είδους πληροφορίες και στατιστική δεν έχουμε, αλλά σίγουρα μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ζώων που μετακινούνται ετησίως από τη μια χώρα μέλος στην άλλη. Τώρα όσον αφορά εθνικό μητρό όλων των σκύλων και το καθεξής, θεωρούμε πως είναι υπερβολική ε, γραφειοκρατία κάτι τέτοιο. Αφόσον ο κανονισμός έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής ε, και τα μοναδικά προβλήματα που έχουμε προκύπτουν από παράνομη εισαγωγή ζώων, δηλαδή πέρα από τους κανόνες εδώ μπαίνουμε σε μια συζήτηση σε σχέση με τους ελέγχους, τους πόρους που δίνονται για ελέγχους, αλλά όχι ακριβώς ε, τα όσα αφορούν αυτό τον κανόνα. Τώρα, για τους εξοδοτημένους ε, κτηνίατρους, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ένα άρθρο, συγκεκριμένα το 18, που αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, διπλώματα των κτηνιάτρων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, εμφύτευση μικροτσίπ. Τώρα αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη αδειοδοτούν τους κτηνίατρους που μπορούν να κάνουν μια ολόκληρη σειρά ε, εγχειρήσεων ας εμβολιασμούς, ε, τοποθέτηση του μικροτσίπ και μετά την έκδοση διαβατηρίου. Ευχαριστώ Κομισιόν προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 27 Ενάτου θα ψηφίσουμε την έκθεση στις 6 Νοεμβρίου και δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα καταλήξει στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμμετοχή στην συζήτηση και προχωρώ τώρα στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι μια ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν για την δηλητηρίαση από μεθανόλη στην τσεχική δημοκρατία. Κάτι που δεν είναι καθαρά εθνικό πρόβλημα της χώρας αυτής, αλλά γιατί έχει σημειωθεί και αλλού. Και εκεί ανέλαβε ο συνάδελφος Πάβελ Ποκ την σχετική πρωτοβουλία και προχωρούμε σήμερα σε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας ακούσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποιο επίπεδο γίνεται κάποια παρέμβαση σε όλη την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια υποστήριξη δίνεται για να ξεκαθαριστεί ας πούμε η κατάσταση. Με συγχωρείτε. Ναι. Α, Πάβελ Ποκ πρώτα. Πάβελ Ποκ και μετά η Κομισιόν. Παύελ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, πρώτη πρώτο περιστατικό δηλητηρίασης από ε, μεθανόλη στην ε, Δημοκρατία της Τσεχίας διαπιστώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου και αυτό μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Ε, υπάρχουν 27 θύματα και πολλά από αυτά βρίσκονται ακόμα στα νοσοκομεία. Οι αρμόδιες αρχές της Τσεχίας αντέδρασαν την περασμένη Παρασκευή. Απαγορεύθηκε η πώληση 20% των ε, αλκοολούχων ποτών με πάνω από 20% περιεκτικότητα σε αλκοόλ και αναζητείται η προέλευση αυτής της μεθανόλης αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να εγγραφεί στο πρόγραμμα της ημερήσία μας διάταξης το θέμα γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την ε, Τσεχία αλλά έχει επηρεάσει και τις γειτονικές μας χώρες πέρα από τα σύνορα. Μήπως τα κράτη-μέλη δεν θα έπρεπε να προχωρήσουν με συντονισμένο τρόπο. Η Πολωνία απαγόρευσε την συμπόληση αλκοόλ τσεχικής προέλευσης, η Σλοβακία το ίδιο, η Γερμανία επίσης σκέφτεται να κάνει το ίδιο. Και θέλω λοιπόν να θέσω την εξή ερώτηση προ την Κομισιόν. Μάλιστα, έχω τρει ερωτήσει να θέσω προ την Κομισιόν, γιατί είναι ερωτήσει κλειδιά κατά τη γνώμη μου. Και είναι σημαντικό, νομίζω, η Επιτροπή μα να ενημερωθεί σωστά, γιατί είναι αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα αρμόδιες τσεχικές αρχές, ποιο είναι το σημείο επαφής, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει μια παρόμοια κατάσταση ώστε να μπορέσει να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα και ποια είναι αυτά τα μέτρα. Για παράδειγμα, η απαγόρευση της πώληση στην τσεχική επικράτεια αλκοόλ ή η απαγορευση εισαγωγής τσεχικού αλκοόλ στις υπόλοιπε χώρες. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία δίνω ευθύ αμέσω το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Στις 10 Σεπτεμβρίου η Τσεχική Δημοκρατία ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για το πρόβλημα αυτό κατανάλωσης μεθανόλης. Οι δηλητηριάσει ε, έχουν ως αποτέλεσμα 23 επιβεβαιωμένους θανάτους και τα τελευταία στοιχεία μιλάνε για 39 άτομα που είναι στο νοσοκομείο, ενώ τα στοιχεία μου έλεγαν για 35. Στην Πολωνία αναφέρθηκαν δύο περιπτώσεις. Στην Σλοβακία 8 ελαφρά δηλητηρίαση. Αυτά γνωρίζουμε. Όλες αυτές τις περιπτώσεις σχετίζονται με κατανάλωση ινοπνεύματος, ινοπνευματοδών που προέρχονταν από την Τσεχία. Στην εσωτερική αγορά όλα τα ενοπληματόδηποτα με πάνω από 30% απαγορεύτηκε στις 13 Σεπτεμβρίου και απαγόρευσε την πώληση όλων των ενοπνευματοδών με πάνω από 20% στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή και άλλα κράτη-μέλη ενημερώθηκαν για αυτά τα εθνικά μέτρα στις 17 μέσω του συστήματος ενημέρωσης. Αυτή η απαγόρευση για όλα τα ενωμένα με πάνω από 20% που εφαρμόζει η Τσεχική Δημοκρατία δεν καλύπτει τις εξαγωγές. Η απαγόρευση αφορά όλα τα ελοπλανατώδη ποτά, όχι μόνο τα τσεχικά. Γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο παραχαραγμένων ετικετών. Το πρόβλημα λοιπόν ακόμη συνδέεται απευθείας με την τσεχική δημοκρατία. Αλλά υπάρχει κίνδυνος λοιπόν εξαγωγής επικίνδυνων, ε, ε, επικίνδυνων ποτών. Και η Πολωνία και η Σλοβακία έχουν πάρει μέτρα προσωρινή απαγόρευση τσεχικών τέτοιων προϊόντων με πάνω από 20%. Αποφασίστηκε αυτός 16% και από χτες και στη Σλοβακία ταυτόσιμη απαγόρευση. Η Κομισιόν επιτηρεί την κατάσταση, λαμβάνει ενημέρωση τακτική από τις αρχές των τριών αυτών χωρών. Από τότε που ενημερώθηκε το σύστημα ταχεία, ταχείας ε, προειδοποίησης. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με τις τρεις χώρες αυτές μέλη. Έχουμε ενημερώσει και άλλα κράτη-μέλη, έχουμε συναντήσεις της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας. Η πρώτη έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη στις 17 Σεπτεμβρίου. όπου ενημερώθηκαν ε, γιατί παρευρίσκονταν οι αρχές των ε, κρατών μελών για τη δημόσια υγεία. Επίσης, η μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων και Υγείας των Ζώων ενημερώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη. και ζητήσαμε ενημέρωση από την Πολωνία και την Τσεχία και το θέμα θα ξαναζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση αυτής της μόνιμης επιτροπής την προσοχή Παρασκευή. Τονίσαμε σε όλες αυτές τις συναντήσεις την ανάγκη έγκαιρης και ορθής ενημέρωσης. Επίσης, η τσεχική κυβέρνηση θα επανεξετάσει τα μέτρα που έχει λάβει σήμερα. Η Επιτροπή ζήτησε τις, από τις τσεχικές αρχές και σε συνάντηση του Κορεπέρ σήμερα το πρωί αλλά και σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη με μεταξύ του ε, Επιτρόπου Ντάλι και του ε, Τσέχου Υπουργού να επεκταθεί αυτή η απαγόρευση και στις εξαγωγές αλκο, ε, από την Τσεχία. Ενημερώσαμε τις τσεχικές αρχές ότι αν τα μέτρα αυτά δεν επεκταθούν και στις εξαγωγές η Επιτροπή θα ε, λάβει τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές στα άλλα κράτη-μέλη και να αποφύγει τη λήψη περαιτέρω μονομερών μέτρων από άλλα κράτη-μέλη. Τη βοήθεια που μπορούμε τώρα να προσφέρουμε στη Τσεχική Δημοκρατία, ο Επίτροπος Ντάλη σήμερα το πρωί, σε αυτήν την τηλεφωνική διάσκεψη με τον Υπουργό, προσέφερε την βοήθειά του χωρίς να διευκρινίσει τι είδους ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν. Αυτό σε τελευταία ανάλυση και σε πρώτη ανάλυση. Βεβαίως ε, είναι θέμα των Τσέχων να ε, εξακριβώσουν και να ε, μας ενημερώσουν για τις ανάγκες τους. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ένας αριθμός συναδέλφων έχουν ήδη εγγραφεί. Και πρώτος ο κύριος Μαστάλκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι Τσέχος ε, Ευρωβουλευτής και βέβαια είμαι και πολίτης και γιατρός και γι' αυτό θεωρώ την κατάσταση αυτή εξαιρετικά δραματική. Έχω την αίσθηση ότι οι αρμόδιες αρχές αντέδρασαν με καθυστέρηση. Διότι θα έπρεπε ήδη να είχαν, να είχαν πληροφορίες ότι διακινείται νοθευμένο ενόπνευμα από τα δίκτυα διανομής και θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει με άλλες μεθόδους και όχι μόνο με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Διότι ως γιατρός θα σας πω ότι αν δεν ασκηθεί έγκαιρα πρόληψη, βέβαια τότε μετά το μόνο που μένει είναι η οδυνηρή καταστολή. Τώρα αυτή η καθυστερημένη αντίδραση έχει ως τραγικές συνέπειες όχι μόνο τους θανάτους και τις, ε, και, τους, και τις νόσους, και τους, δηλαδή τους ανθρώπους που βρίσκονται στα νοσοκομεία, αλλά και προβλήματα στην διακίνηση εμπορευμάτων. Πρέπει να δει τώρα η Τσεχική Δημοκρατία τι μπορεί να κάνει για να σταματήσει τις ε, εξαγωγές αυτές, καθώς επίσης να επιβάλλει και τις απαραίτητες κυρώσεις σε αυτούς που δεν έπραξαν το καθήκον τους. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργαζόμαστε έκθεση για τις νέες απειλές κατά της υγείας του κοινού και στα πλαίσια αυτά βέβαια καλούμαστε να επισημάνουμε τις νέες απειλές. Όλα αυτά βέβαια είναι ε, πολύ σημαντικά πράγματα, είναι ωστόσο και δαπανηρά. Και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο η τσεχική πλευρά ήταν ενήμερη για το πρόβλημα και τι αναμένει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξουν οι τσεχικές αρχές. Děkuji. Αγαπητοί συνάδελφοι, η καταστροφή, και το λέω καταστροφή, δεν είναι πολύ να το πούμε αυτό, έχει δραματικές επιπτώσεις σε όλη τη χώρα, και σε τόσες δεκάδες άτομα και οικογένειες και οικονομικές επιπτώσεις έχουμε αλλά και διεθνείς επιπτώσεις, διεθνούς επίπεδου. Τονίζω ότι είναι μια εντελώ ασυνήθιστη κατάσταση που ουδέποτε είχε προκύψει στη χώρα μας. Ποτέ δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ε, κρίση. Αλλά έχουμε και άλλες εμπειρίες από την Εστονία το 2001 όπως και εκεί, γιατί όταν και εκεί προέκυψε πρόβλημα δηλητηρίας από μεθανόλη, υπήρξαν θάνατοι, ή στην Νορβηγία 2004 πέθαναν 59 άτομα από τέτοια δηλητηρίαση. Ο Λέος ο Τσέχος Υπουργός Υγείας, με ενημέρωσε και θα ήθελα να σας πω ορισμένα από αυτά που μου είπε. Σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνησή μας αντέδρασε πολύ γρήγορα, όπως αναφέρθηκε ήδη, στις 12 Σεπτεμβρίου. Απαγορεύτηκε η πώληση σε καταστήματα, από καταστήματα και από κιόσκια ε, και κατόπιν γενικότερα όλων των ινοπνευματοδών με πάνω από 20%. Η χώρα μου εισήγαγε μια σειρά ε, τα τελευταία χρόνια μέτρων για έλεγχο. Το 2011 έγιναν πάνω από 40.000 έλεγχοι και την προηγούμενη χρονιά έγιναν πολύ δειγματοληπτικοί έλεγχοι και παρά τις τόσες δεκάδες χιλιάδες ελέγχους ποτέ δεν είχαμε διαπιστώσει περιεκτικότητα μεθανόλης στα ποτά αυτά. Οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για μεθανόλη που εισήχθη συμπληρωματικά στο ποτό. Όχι ε, μεθανόλη η οποία δημιουργείται κατά τη διάρκεια απόσταξης ε, κατασκευής του, των ποτών αυτών. Αυτό που και μένα με εξέπληξε είναι τι υψηλό, υψηλή περιεκτικότητα μεθανόλης ήταν το 2009 στην Τσεχία εισήχθησαν πάνω, 10, πάνω από 10 τόνους μεθανόλης από τη Γερμανία και από τη Ρωσία. Είναι λοιπόν δυσχερές και περίπλοκο το πρόβλημα αυτό και μια πλευρά του ζητήματος έχει να κάνει με την διεθνή φήμη και υπόλοιψη της χώρας μου. Πρέπει οπωσδήποτε να επιλύσουμε σύντομα το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει ενεργητική επικοινωνιακή πολιτική. Πρέπει να παρέχεται με διαφάνεια η τελευταία πληροφόρηση σε όλους, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τραγικό πρόβλημα. Τρεις ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Ήδη τις αναφέρατε εν μέρη. Θα ήθελα να μάθω μέχρι τώρα και στο μέλλον πώς ε, θα σχεδιάσετε την ε, συνεργασία μεταξύ Κομισιών Τσεχίας και άλλων κρατών μελών, τι οδούς θα ακολουθήσει, πώς η Κομισιόν θα βοηθήσει την Τσεχία και τις άλλες χώρες. Και τρίτον, τι διδάγματα μπορούμε να εξαγάγουμε από αυτή την ε, κρίση μεθανόλης, τι προγράμματα μπορούμε να εισαγάγουμε στο μέλλον και μέσω της Επιτροπής μας. Να δώσω τώρα το λόγο στην προηγούμενη, στην πρώτερη ε, Υπουργό ε, Υγείας της Τσεχικής Δημοκρατίας, την κυρία Χόιτεβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θεωρώ την κατάσταση αυτή ως πραγματική καταστροφή διότι υπήρξαν ανθρώπινα θύματα και Ίσως μάλιστα να προσθεθούν και άλλοι θάνατοι τώρα από τα πρόσωπα που νοσηλεύονται. Δεν πρόκειται μόνο για την κατάσταση στην τσεχική δημοκρατία, αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινού στην ενιαία αγορά. Η τσεχική κυβέρνηση αντέδρασε με τρόπο διαφανή από την αρχή και διέθεσε τις πληροφορίες που γνώριζε και στους εταιρούς της αλλά και στην κοινή γνώμη και βεβαίως συνεργάστηκαν διεθνώς οι αρμόδιες αρχές. Εγώ είμαι ικανοποιημένη διότι λειτουργήσε καλά το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση της Ένωσης και το Τσεχικό Υπουργείο διαβίβασε με ταχύ τρόπο τις πληροφορίε που διέθετε. Θέλω να κάνω ωστόσο μια διόρθωση. Λέχθηκε προηγουμένως ότι διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες στις 9 Σεπτεμβρίου. Αλλά εγώ ε, γνωρίζω ότι ήταν ήδη νωρίτερα και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Τσεχή Δημοκρατία έπραξε παν το δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι το ενόπνευμα αυτό δεν θα καταλήξει στο εμπόριο. Τώρα υπάρχουν προτάσεις τα μπουκάλια που περιέχουν ενοπνευματώδη ποτά να συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό προέλευση τους. Το ερώτημα είναι βέβαια πώς θα εξασφαλιστεί βέβαια και το εμπόριο μέσω του διαδικτύου. Ο κύριος Ποκ διαβίβασε στην Προεδρία της Επιτροπής μας επιστολή με τις σχετικές πληροφορίες και εδώ οφείλω και να κάνω μια δεύτερη διόρθωση. Ένα μέρος του τσεχικού κοινού, και αυτό είναι βέβαια ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα μειονεκτικών περιφερειών, έχει την εντύπωση ότι παραμελείται από την κυβέρνησή του. Και γι' αυτό ε, λέει η επιστολή ότι είναι καλό να επιληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ε, θα ήθελα να αποστασιοποιηθώ από αυτή την δήλωση του συναδέλφου μου κ. Ποκ η ποτσ Θεωρώ ότι αυτά ε, τα λέει διότι σε ένα μήνα επίκειται οι περιφερειακές εκλογές και εν ώψη αυτών προσπαθεί να ρίξει το πολιτικό φταίξιμο σε άλλους. Νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι σωστή. Η κυρία Ροτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ να προσπαθήσουμε να αφήσουμε εκτός την ε, υπόθεση αυτή της ο κ. Καμπρνός δεν έχει μετάφραση. Ε, θα τα πω στα αγγλικά τότε. Ξαναλέω λοιπόν, λέει η Δάγμα Ροτπέρεντ, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε απ' έξω τους ενδοτσεχικούς καυγάδες ε, πολιτικής μορφής. Σας τα αφήσουμε απ' έξω. Οι συνάδελφοι που είναι παρούσες και παρόντες θα συμφωνήσουν ότι ήταν σωστό το μέτρο και η πράξη του κυρίου Πότς που τα έθεσε υπόψη μας. Όλοι θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Και εγώ το ίδιο. Εγώ δεν το σκέφτηκα, το ομολογώ. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον συναδελφό μα. γιατί καθήκον μα είναι να εγγύψουμε στο θέμα αυτό. Μιλάμε για νοθευμένα φάρμακα, μιλάμε για παντίους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και εδώ είναι κάτι το οποίο είναι, ε, θα έπρεπε να είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας. Για μένα είναι σαφές ότι εδώ από πίσω κρύβονται εγκληματικές διαθέσεις, τι οποίες βέβαια δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε. Είναι σαφές ότι εγκληματίε οι οποίοι αποβλέπουν στο να βλάψουν άλλους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο να αποτραπούν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα πυκνό δίχτυ ελέγχων ως αποτροπή. Εγώ παρακολουθώ τις σχετικές δημοσίευσεις ό,τι βλέπω δηλαδή σε γερμανικά και αγγλικά μέσα, γλώσσες που καταλαβαίνω τέλο πάντων, τα διάβασα όλα αυτά και βρήκα σωστό ότι αμέσως επιβλήθηκε απαγόρευση διάθεση στο εμπόριο υνοπνευματοδών με περιεκτικότητα άνω του 20% συνόπνευμα. Δεν είμαι απόλυτα βεβαία και συμφωνώ με τον κύριο Μαστάλκα, για το πόσο γρήγορα αντέδρασε η τσεχική κυβέρνηση, γιατί εδώ μετράνε οι ώρες. Άκουσα προσεκτικά και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, που εντάξει λειτουργεί το σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης εφόσον μια χώρα δηλώνει το συμβάν. Χαίρομαι και που συζητήθηκε και ε, στου μονίμου αντιπροσώπου ότι ο κύριο Ντάλι πήρε τηλέφωνο τον Τσέχο Πρωθυπουργό. Όλα αυτά καλά είναι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι δύο πράγματα. Αφενός θα ήθελα ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, να γνωρίζω πότε έγινε γνωστή η πρώτη περίπτωση στην Τσεχία. Δηλαδή, τη δήλωση κάποιου γιατρό, στο νοσοκομείο, πότε επέβαλε την απαγόρευση η τσεχική κυβέρνηση και δεύτερον η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε ενημερώθηκε στα πλαίσια του Rapid Alert. Νομίζω αυτό πρέπει να γίνεται 48 ώρες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε εδώ. Και θέλω ακόμη να γνωρίζω ο κύριος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα όταν δεν είναι σίγουρο ότι απαγορεύεται το εξωτερικό εμπόριο. Άρα δηλαδή ότι τίποτε δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει την τσεχική επικράτεια. Εσείς διευκρινίσατε τα μέτρα αυτά με την τσεχική κυβέρνηση και τι προτίθεστε να κάνετε, πότε θα λάβετε αυτά τα μέτρα προφύλαξης. Γιατί μου φαίνεται σωστό που έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει, δεν είμαι βεβαία ότι πράγματι κινήθηκαν όλοι με την ταχύτητα που έπρεπε, Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται, όπως άλλωστε και με την όθευση φαρμάκων, φαίνεται ότι αυτή η εγκληματική διάθεση επιτρέπει τελικά την όθευση με τοξικές ουσίες, ποτών και άλλων καταναλωτικών ειδών, και πρέπει να μάθει η Κομισιόν από την τσεχική κυβέρνηση με ποιον τρόπο προτίθεται να αναζητήσει την πηγή του κακού. το λέω επίτηδες προσπαθήσει, διότι δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια. Και πώς λοιπόν θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πάβελ Κότς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κομισιόν απάντησε στα ερωτήματά μου Ευχαριστώ για την βοήθεια που προσέφερε, από ό,τι κατάλαβα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η πρέπουσα βοήθεια προς την τσεχική βοήθεια, προς την τσεχική δημοκρατία όταν ζητηθεί. Τον ευχαριστώ. Ήταν ε, σημαντικό και καλό που το άκουσα αυτό, που το είπε αυτό. Δεύτερο, και νομίζω ότι είναι η κοινή μας άποψη όλων των μελών της Επιτροπής, είναι σημαντικό να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας ε, στους συγγενείς των θυμάτων, την συμπαράστασή μας ε, στους ασθενείς στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό εκ μέρους όλων. Να εκφράσουμε τη λύπη μας. Κατά τα άλλα, τα άλλα θέματα, τα μικροπολιτικά τα αφήνω. Ετέθησαν κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε παρακαλώ και την Κομισιόν να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τώρα την διαδοχή των γεγονότων. στις 10 Σεπτεμβρίου πήρε μέσω του Rapid Alert την ειδοποίηση. Η Τσεχία, να διορθώσω, στις 8 Σεπτεμβρίου εισήγαγε ως πληροφόρηση στο σύστημα αυτό Rapid Alert τα στοιχεία αυτά. Οπότε δεν ε, ε, ελήφθη αμέσως μέσω του συστήματος ως αίτιο συναγερμού. Είχαν γίνει κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις 6 Σεπτεμβρίου. Έτσι λέει μέσα στο σύστημα η ενημέρωση. Μπορώ να αναφέρω μόνο την ενημέρωση όπως είναι μέσα στο σύστημα αυτό ταχαίου συναγερμού. Rapid alert. Κατόπιν Όπως ήδη είπα, στις 10 Σεπτεμβρίου λάβαμε αυτόν, αυτόν τον συναγερμό και κάναμε μία πρώτη ενημερωτική συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους κρατών μελών στις 13 ε, ε, στην μόνιμη επιτροπή για την επιστηστική ασφάλεια, ασφάλεια τροφίμων. Συμμετείχαν και εκπρόσωποι από τις τρεις ε, βεβαίως θυγόμενες χώρες. Για τα ερωτήματα της κυρίας Ροτ Μπέρεντ. Εάν διευκρίνησε έναντι της Κομισιόν τα μέτρα η Κομισιόν, Εάν η Κομισιόν έναντι της Τσεχίας διευκρίνησε τα μέτρα, τους είπα λοιπόν ότι όλα τα ενοπνευματώδη με πάνω από 20% απαγορεύτηκαν στην Τσεχία. Όλα τα ενοπνευματώδη ανεξάρτητα από, τύπου, από τύπο ή προέλευση. η Σλοβακία και η Πολωνία έλαβαν ανάλογα μέτρα για εισαγωγές συνοπληματοδών από την Τσεχία. Ο Επίτροπος Ντάλιν διευκρίνησε σήμερα στον Τσέχο Υπουργό ότι αν τα μέτρα δεν ε, επεκταθούν και για προϊόντα που εξάγονται σε άλλες χώρες μέλη θα λάβει μέτρα η Κομισιόν. Δεν διευκρινίσαμε και δεν ήμασταν σε θέση να το κάνουμε όπως υπόθηκε ο ενδεχόμενος περιορισμός των υνοπνευματοδών ε, με βάση την πληροφόρηση που έχουμε ως τώρα δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποια είναι ο αφορά. Δεν έχουμε καμία εγγύηση εάν μπορούμε να εξαιρέσουμε κάποια εινοπνευματόδη από αυτήν την απαγόρευση. Οπότε ισχύει για όλα τα ποτά η απαγόρευση. Και αν δεν υπάρξει απαγόρευση εξαγωγών, η Κομισιόν θα εισαγάγει ταυτόσημα με τα τσεχικά μέτρα σε επίπεδο ένωσης. Θα απαγορεύσει την εξαγωγή όλων των υλοπηματοδών σε κοινοτικό επίπεδο. Προέλευση αυτών των ποτών. Δηλαδή ποιο έκανε αυτές τις εγκληματικέ πράξεις. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει αστυνομική έρευνα. Αυτό είναι θέμα ελέγχων, είναι θέμα αστυνομίας. Δεν έχουμε καμία περαιτέρω πληροφόρηση. δεν μπορώ να βοηθήσω, οι αρμοδιότητες μου δεν με επιτρέπουν να βοηθήσω την αστυνομία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και πλαστές ετικέτες σε αυτά τα μπουκάλια διαφόρων ειδών ίνοπνευματοδών. Όσες τέτοιες πλαστές ετικέτες έχουν βρεθεί, έχουν γίνει δημοσίως γνωστές, αλλά η πηγή αυτή καθεαυτή ως τώρα δεν είναι γνωστή. Τι βοήθεια τώρα μπορούμε να δώσουμε. Όπως είπα, προσέφερε ο Επίτροπος Ντάλι. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα τι μορφή θα λάβει αυτή η βοήθεια, θα μπορούσε να λάβει. Θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία της εικόνας. Μπορούμε να βοηθήσουμε με εργαστηριακές αναλύσεις, Δεν έχω συγκεκριμένα προγράμματα, σχέδια αυτή τη στιγμή για το τι είδος βοήθειας πρέπει να διευκρινίσει και η τσεχική πλευρά. Πρόεδρος. Δεν έχω τι να πω. Και άλλοι συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Πρώτα η συνάδελφος Ροτ Μπέραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε τη λειτουργία του συστήματος Rapid Alert σε σχέση με προβλήματα με τρόφιμα. Πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά καταπληκτική κατάσταση. Εντάξει. Δεν θα πιω πλέον ε, τέτοιου είδους ποτά. Έχω δύο παρακλήσεις. Έχουμε αρκετά σαφείς κανόνες στην Ένωση πώς πρέπει να κυκλοφορεί η ενημέρωση από το ένα κράτος μέλος προς τα άλλα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με τα τρόφιμα όταν υπάρχουν προβλήματα με, ε, νόθευσης στις 6 λοιπόν Σεπτεμβρίου διαπιστώσαμε το πρώτο πρόβλημα με τη μεθανόλη. Τα στοιχεία αυτά τα έβαλε η Τσεχία στις 8 ενάτου και εσείς τα λάβατε στις 10 ενάτου. Έχουμε πρόβλημα. Να ρωτήσουμε τους Τσέχους λοιπόν τι έκανε ακριβώς στην πράξη. Επιπλέον, απόλυτα σωστό είναι το ότι τα ενοπνευματόδη με άνω 20% απαγορεύτηκε να πολλούνται. Αλλά νομίζω ότι είναι κοινικό να πούμε. Δεν τα πουλάμε στη χώρα μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά οτιδήποτε είναι για εξαγωγή και ενδεχομένως είναι επικίνδυνο, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Το ότι δεν ε, απαγορεύτηκαν και οι εξαγωγές δεν το καταλαβαίνω. Ίσως να, διανοητικά να μην είμαι επαρκή, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Στις 13 ενάτου έγινε μια συνεδρίαση, ωραία, θαυμάσια. Ο χρόνος που πέρασε, 10 ελάβατε την ενημέρωση, 13 Ενάτου. Θα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί τα μέτρα διασφάλισης. Και σήμερα έχουμε ακόμη 19. Και σήμερα μίλησε ο κύριος Ντάλι με τον Υπουργό. Πρέπει να έχετε την εγγύηση ότι αύριο θα σταματήσουν οι εξαγωγές. Τότε, εάν δεν ε, έχετε αυτή την ε, εγγύηση, θα πρέπει να λάβετε εσεί τα μέτρα διασφάλισης. Πώς θα εξηγήσετε στο ευρωπαϊκό κοινό ότι οποιοδήποτε αγοράσει ένα μπουκάλι ε, ποτό, δεν ξέρω πού, στη Δανία, θα του πούμε, θα το πούμε αν πάθει μετά κάτι, με συγχωρείτε, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά είναι επικίνδυνα για τη ζωή την ίδια των ανθρώπων. Παίζουμε ρωσική ρουλέτα. Τι μπουκάλι έχω. Είναι επικίνδυνο ή όχι, γιατί δεν έχουμε βρει την πηγή. Δεν ξέρω ποιο φέρει την ευθύνη. Δεν θα ήθελα εγώ να τη φέρω. Και θα ήθελα να σα καλέσω εσά και στον κύριο Ντάλι, που είναι υπεύθυνο, να προσέξει να μην τη φέρει εκείνο αυτή την ευθύνη. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μαστάλκα. Και μετά η Τιότοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια συμπληρωματική ερώτηση μετά τα όσα άκουσα από την ε, Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για ενδοτσεχικούς καυγάδες πριν από τις εκλογές. Έχουμε μιλήσει για ε, προθέσεις ε, που χρησιμοποιούνται μετά από επεμβάσεις, έχουμε μιλήσει για το φάρμακο Mediator και ούτω καθεξής. Άλλο ένα, θέμα, άλλο ένα τέτοιο σκάνδαλο είναι. Έχω λοιπόν μια ερώτηση προς την Κομισιόν για δική μου πληροφόρηση. Ποια είναι η διαφορά κατά τη γνώμη σας μεταξύ δηλώσεως, μεταξύ εισαγωγής της πληροφορίας στο σύστημα Rapid Alert στις 8 και της άφηξής του σε εσά στις 10. Τι συνέβη. Υπήρξε κάποιο σφάλμα. Όχι απαραίτητα δηλαδή από την τσεχική δημοκρατία. Ίσως υπάρχει κάπου κάποιο πρόβλημα, κάποια έλλειψη. Επίσης, συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφό μου για την έκφραση συλληπιτηρίων. Εγώ βέβαια είμαι αναπληρωματικό μέλο, αλλά επιθυμώ να συμμετάσχω στην έκφραση συλληπιτηρίων. Η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στη χρονολογική σειρά των γεγονότων. Στις 6 Ενάτου σημειώθηκαν δύο θάνατοι, οι οποίοι κατανάλωσαν ενόπνευμα το, αγόρα, το οποίο αγόρασαν στον δρόμο. Η αυτοψία κατέδειξε ότι επρόκειτο για δηλητηρίαση από μεθανόλη και μετά σημειώθηκαν και άλλοι θάνατοι στην ίδια περιοχή. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης να δηλωθεί ο κάθε θάνατος που μπορεί να ε, συμβαίνει από τέτοια πράγματα. Μόνο όταν διαπιστώνεται από τον αριθμό των θανάτων και από άλλα στοιχεία ότι πρόκειται για ένα ενδεχόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας, δηλαδή ευρύτερο. Μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η μεθανόλη ε, φτάνει στο τελικό προϊόν λόγω της απόσταξης που γίνεται με παράνομους τρόπους κατοίκων κτλ. Μετά με την αυτοψία διαπιστώθηκε περί τίνος επρόκειτο και λήφθηκαν απαραίτητα μέτρα και έγινε τότε και η εισαγωγή της πληροφορίας στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Σχετικά με τις πηγές τώρα, υπάρχουν καμιά φορά και εσφαλμένες πληροφορίες. Έχει σημειωθεί και άλλη παλαιότερη περίπτωση με μόλυνση που προήλθε από άγνωστες πηγές. Και σημαντικό είναι, ιδίω για την ενιαία αγορά, τα μέτρα να είναι επίσης προσαρμοσμένα και αναλογικά. Και γι' αυτό χαίρομαι που η Κομισιόν επιθυμεί να υποστηρίξει την τσεχική δημοκρατία στην λήψη των μέτρων για να φροντίσει ώστε αυτά να είναι πραγματικά ανάλογα. Ε, υπόκειται δηλαδή στην αρχή της αναλογικότητας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η, η ερώτηση μου δεν απαντήθηκε. Και εννοώ την οδηγία για διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Θα ήθελα εδώ να ακούσω ποια διδάγματα αντλείται από την υπόθεση αυτή. Είναι σημαντικό που λάβαμε τις πληροφορίες και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, αλλά δεν είμαστε όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Θα ήθελα να μάθουμε ποια είναι τα διδάγματα τα οποία αντλεί η Κομισιόν από την υπόθεση αυτή για να προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα και για να μπορέσουν βέβαια να διατυπωθούν οι κατάλληλες προτάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιοι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στο μέλλον και να βελτιωθεί το σύστημα. Υπάρχει νομοθεσία που είναι βέβαια το Rapid Alert System, λέει ο πρόεδρος, για food και feed, δηλαδή για τρόφιμα και ζωοτροφές και εκπλήσωμε ακόμα από το κενό που διαπιστώνουμε ανάμεσα στην δήλωση στο σύστημα μέχρι τη στιγμή που ήλθε. Βέβαια είναι το Σαββατοκύριακο στη μέση. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά πώς είναι δυνατόν να προκύψει τέτοια καθυστέρηση. Εκεί τα λεπτά και οι ώρες έχουν κρίσιμη σημασία, είναι αποφασιστικά. Ας θέσουμε το θέμα αυτό υπόψη των συντονιστών, αν ίσως πρέπει να το διαφωτίσουμε περισσότερο. Γιατί όπως λέω, κάθε λεπτό που περνάει και κάθε ώρα που περνάει έχει τεράστιο κόστος. Εδώ έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι. Και σε ό,τι αφορά την απαγόρευση εξαγωγών, νομίζω λέχθηκαν αρκετά γι' αυτό. Θα δώσω το λόγο πάλι στην Κομισιόν για να απαντήσει και να απαντήσει σε όσα άλλα μπορεί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως υπόθηκε, στις 6 Σεπτεμβρίου έγιναν κάποιοι δειγματοληκτικοί έλεγχοι. Η εισαγωγή στο σύστημα έγινε στις 8. Αυτό έχει να κάνει με το ότι τα δείγματα λήφθηκαν στις 6. Πρέπει πρώτα απ' όλα όμως τα δείγματα αυτά να εξεταστούν, να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Τσεχική Δημοκρατία ότι πρέπει να γίνει εξέταση των δειγμάτων. Στις 8 εισήχθησαν και στις 10 έφτασαν στην Κομισιόν. Έτσι έχουν τα πράγματα. τι διδάγματα μπορούμε να εξαγάγουμε. Όσο δεν έχει διαλευκανθεί η υπόθεση, όσο δεν ξέρουμε πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα, αν είναι οργανωμένο, αν είναι μεμονωμένο, δεν μπορώ να εκφραστώ. Είναι ένα θέμα μεγάλων διαστάσεων που δεν είναι δικό μου θέμα να το απαντήσω. Είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης ε, άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε στο μέλλον να προλαμβάνουμε τέτοια κρούσματα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα της ε, υπόθεσης. Δεν έχω σημειώσει καμιά άλλη ερώτηση προς εμένα. Με συγχωρείτε αν ε, δεν απάντησα σε κάτι. Πρόεδρος. Ωραία. Κλείνουμε την συζήτηση ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θλιβερό γεγονός για άλλη μια φορά να εκφράσω τη συμπάθειά μου, τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων και θα γίνει και με γραπτή μορφή. Πρέπει να δούμε τι αδυναμίες έχει το σύστημα και γι' αυτό πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Πότς που ζήτησε να εισαχθεί στην ημέρηση διάταξη. Ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το θέμα και για μένα. Εξήγαγα πολλά διδάγματα και εγώ προσωπικά και ελπίζω ότι η Κομισιόν θα κάνει όλα όσα πρέπει για να περιορίσει τι επιπτώσεις αυτής της περίπτωσης, να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα που θα έχουν προβλήματα με την υγεία και με τη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Οπότε εδώ πρέπει να πας, ε, πρέπει να κλείσουμε την ε, συνεδρίασή μας και αύριο στις 9 έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ.